Αγαπητοί συναδελφοί, μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών, παρακαλώ καθίστε για να αρχίσει η συνεδρίασή μας. La Κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεώς μας. Χαιρετίζω την Αντιπρόεδρο Κεργίεβα εδώ, η οποία έρχεται στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, για να μας παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού 2017, έτσι όπως εγκρίθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Αντιπρόεδρε. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για τέσσερις ώρες για τις συνθήκες υποδοχής των προσφύγων και για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ακούσαμε λόγια από τον Τζόρτζο ε, Σόρο στην αρχή που κάποιοι μπορεί να τα κρίνουν ως προκλητικά. Αλλά είπε τι μέσα πρέπει να κινητοποιήσουμε αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πρόκληση αυτή που είναι μια πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Αναφέρθηκε σε 30 δισεκατομμύρια για την χρηματοδότηση είτε με ίδιους πόρους είτε με έναν φόρο επί των καυσίμων, κατανάλωση καυσίμων είτε με δάνεια. Δεδομένου ότι σήμερα τα επιτόκια είναι κοντά στο μηδέν και μερικές φορές και αρνητικά. Συζητήσαμε λοιπόν για τις κατηγορίες 3 και 4, γιατί η κυρία Καλβίνιο ήρθε και συμμετείχε στη συζήτησή μας σήμερα το πρωί και μας παρουσίασε κάποιες πρώτες πληροφορίες που ίσως επιβεβαιωθούν τελικά από το Σώμα των Επιτρόπων. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργίβα που είσαστε εδώ και σας δίνω και τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού σήμερα το πρωί στις 9.30. Είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένη που είμαι παρούσα ήδη σήμερα εδώ ενώπιον σας. Ε, η παρουσίασή μου είναι στα αγγλικά και γι' αυτό συνεχίσω στη γλώσσα αυτή. Εμείς ευχαρίστως δεχόμαστε τους Άγγλους και τα αγγλικά, λέει ο Πρόεδρος. Εδώ. Για τη γλώσσα βέβαια δεν υπάρχει πρόβλημα, δε, κύριε Γεωργίου. Ίσως για τους Άγγλους. Ευχαριστώ λοιπόν. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ε, συναντώμεθα έχει υποστεί τις σημαντικές επιπτώσεις της εκβάσεως του Βρετανικού Δημοσιοφίσματος. Βέβαια, όσον αφορά το έργο μας για τον προϋπολογισμό, δεν έχουμε άμεσες επιπτώσεις από το δημοψήφισμα πέραν της ανάγκης να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από ποτέ τον προϋπολογισμό μας ως ζώνη προστασίας κατά της κρίσεως ως πηγή αναζωογόνησης της ε, απασχόλησης, ε, της ανάπτυξης, ως μια συλλογική προσπάθεια για να ενισχύσουμε τις χώρες μέλη μας που αντιμετωπίζουν μια τεράστια κρίση. Από την αρχή επιθυμώ να δηλώσω ότι συνεχίσαμε με μεγάλη υποστήριξη από το Κοινοβουλίο να κατευθύνουμε τον προϋπολογισμό προς ξεκάθαρες προτεραιότητες και να χρησιμοποιούμε την ευελιξία που μας έχετε χορηγήσει για να προσαρμοστούμε στις ε, περιστάσεις που αλλάζουν. Στη σημερινή μου παρουσίαση θα εγκύψω στα εξής ερωτήματα. Πρώτο, διαφάνεια παρακαλώ. Πρώτα, την τεχνική προσαρμογή που έχουμε λάβει εντολή να εφαρμόσουμε. Δεύτερο, να εντάξω το σχέδιο προπολογισμού στο πολιετέ πλαίσιο. Τρίτο, μια συνολική επισκόπηση υποχρώσεων και πληρωμών. Τέταρτο, δύο προτεραιότητες για το σχέδιο προπολογισμού του 2017, δηλαδή δουλειέ, ανάπτυξη, επενδύσει και από την άλλη μεριά μετανάστευση, προσφυγικό κλπ. Πέμπτο, διοικητικέ δαπάνες και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που έχει σχέση με την ασφάλεια και τέλος την αυξανόμενη σημασία της προσοχής πρέπει να δίδεται στην αποτελεσματικότητα. Ας αρχίσω με την τεχνική προσαρμογή. Όσο θα γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει από τον κανονισμό του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου την εξουσία να κάνει τις τεχνικές προσαρμογές χωρίς να χρειάζεται νομοθετική διαδικασία. Είναι ιδιαίτερο το φετινό έτος διότι πρέπει να περιλάβουμε την προσαρμογή της, ε, των φακέλων της πολιτικής συνοχής που οδηγεί σε μια συνολική αύξηση της τάξης των 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί σε σημερινές τιμές στα 4 δισεκατομμύρια που είχαν πει ως οροφή στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό για τα έτη 2017 2020. Εδώ υπάρχουν τρεις βασικοί δικαιούχοι της προσαρμογής, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, συν πέντε χώρες μέλη, των οποίων θα μειωθούν τα χρήματα που λαμβάνουν, χωρίς όμως κανένα να ξεπερνά, καμία από τις αυτές να ξεπερνά το, 100 εκατομμύρια ευρώ. επιθυμούμε να εστιάσουμε στα πρόσθετα κονδύλια που θα πάνε στις τρεις χώρες που ανέφερα, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, για μετανάστευση, ε, απασχόληση των νέων και επενδύσεις, σε συνεργασία βέβαια με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο μάλλον Στρατηγικών Επενδύσεων. Το σχέδιο προπολογισμού για το 2017 μέσα στο ε, πολιετές πλαίσιο. Το γράφημα που βλέπετε ε, δείχνει δύο, μάλλον δίνει δύο σημαντικά μηνύματα. Ένα, ότι χρησιμοποιούμε πλήρως τον προπολογισμό. Δεν αποτελεί εξαίρεση ο προπολογισμό του 2014. Εάν συγκρίνεται την ανάπτυξη του προπολογισμού τώρα σε σχέση με παλαιότερες περιόδους θα δείτε ότι η προβολή που γίνεται και η χρήση που γίνεται συμπίπτουν. Δεύτερο, στην ε, περίπτωση των υποχρεώσεων βλέπουμε το γράφημα να υπερβαίνει την οροφή διότι το flexibility instrument για τις υποχρώσεις είναι πάνω από την οροφή και έχουμε το μήνυμα για τον προϋπολογισμό του 2017 ότι σε ό,τι αφορά τις πληρωμές η καθυστέρηση για την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων μας αναγκάζει να ζητήσουμε σημαντικά λιγότερα χρήματα. Δηλαδή 6,2% λιγότερα από πέρσι για πιστώσεις πληρωμών. Αυτός είναι πραγματικός λόγος ανησυχίας πρέπει να βρούμε τρόπο όλοι συλλογικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και διότι δεν θέλουμε αυτό το γιο-γιο να αρχίσει, ε, δηλαδή να λειτουργεί στο τέλος της δημοσιονομικής προοπτικής. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει σε νούμερα τον, ε, το σχέδιο προϋπολογισμού. Δεν θα σας βασανίσω ε, διεξερχόμενη γραμμή προς γραμμή αλλά θα έρθω μόνο στις επικεφαλίδες. Συνολικά είναι 75,5%, 157,7% συγγνώμη, για τις υποχρώσεις, 134,9% για τις πληρωμές και τα ποσοστά δίπλα είναι σε σύγκριση με το προϋπολογισμό του 2016 συν 4,7% στις υποχρεώσεις, όμως να μην λησμονήσουμε ότι αυτό απηχεί και τα 21 δισεκατομμύρια σε υποχρώσεις που χρειάστηκε να προτάξουμε λόγω του ότι άρχισε αργά το τρέχον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή στην πραγματικότητα με ονομαστικούς όρους είναι 1,7% η αύξηση και το ποσοστό που ανέφερα προηγουμένως των πληρωμών που μειώνονται κατά 6,2% απέναντι στο, στον προπολισμό του 2016. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω μια συνολικότερη επισκόπηση με ε, γραφήματα που είναι πιο εύκολο να τα δείτε από ένα πίνακα και το πρώτο γράφημα δείχνει την κίνηση προς τα πάνω των υποχρώσεων και προς τα κάτω των πληρωμών. Τα καλά νέα, ωστόσο, για τις υποχρώσεις είναι, όπως θα δείτε αργότερα στην παρουσίασή μου, ότι ευθυγραμμίζουμε την αύξηση με τις προτεραιότητές μας. Τα καλά νέα τώρα για τις πληρωμές είναι ότι μπορούμε να πούμε τώρα ότι τα καθυστερούμενα, εκείνο το backlog από την προηγούμενη δημοσιονομική προοπτική, έχει μειωθεί. Δεν υπάρχει. Δεν φέρουμε, δεν κουβαλάμε πλέον αυτή την ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, μας ανησυχεί η μείωση της ταχύτητας της εφαρμογής νέων προγραμμάτων. Και δεν μπορώ να το επαναλάβω αρκετά για να σας πω δηλαδή πόσο πολύ ανησυχούμε από αυτό. Ας δούμε τώρα το βασικό μήνυμα του σχεδίου προϋπολογισμού. Πολύ στενή ευθυγράμμιση του που πηγαίνουν τα χρήματα με τις προτεραιότητες που έχει στηρίξει το Κοινοβούλιο. Αύξηση της απασχολήσεως, επενδύσεις, αποτελεσματική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση προσφυγικού μεταναστευτικού και όπως είπε και ο πρόεδρος σας Αρτουή, σας έδωσε ήδη και μια ιδέα το πώς θα εξελιχθούν οι προτεραιότητες για το 2017. Βάζουμε τον προϋπολογισμό αυτό στα πλαίσια της αναζήτησης αποτελεσμάτων και πολύ πιο ρητά και ξεκάθαρα στοχεύουμε στην performance, στην απόδοση. Όχι μόνο πόσα χρήματα που, αλλά για και πώς θα γνωρίζουμε αν πραγματικά ο προπολογισμό χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν εξετάσετε τώρα την επόμενη διαφάνεια για δουλειές, ανάπτυξη και επενδύσεις, θα δείτε εδώ ότι έχουμε μια συνολική αύξηση 11% στον τίτλο 1α, αύξηση η οποία φτάνει σε κάθε μέρος το 1α. Για το ευσύ, όπως σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε από όλους μας 29,5, για το Horizon 2020 συν 7,9, για τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη 14,7%, για το Ερασμό συν 16,2% και το συνολικό απόλυτο ποσό είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, παραπάνω που διοχετεύονται σε τομείς προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να τονίσω ότι εξελίσσεται όπως είχαμε συμφωνήσει, έχουμε δημιουργήσει μέσα σε ένα χρόνο για το ΕΦΣΥ η δηλαδή. Είχαμε βάλει περίπου το 1 τρίτο των συνολικών επενδύσεων και είμαι πολύ ευχαριστημένη διότι τα πάμε καλύτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ταχύτητα με την οποία χρησιμοποιούμε το τμήμα εκείνο που προορίζεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του EFSI είναι τόσο καλό πρέπει να βρούμε, τόσο ταχύ, ο πρέπει να βρούμε τρόπους να το ενισχύσουμε. Γιατί, διότι γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνε που παράγουν απασχόληση και αυτό θέλουμε στην οικονομία μας. Αν εξετάσετε τώρα την επόμενη διαφάνεια που δείχνει τι γίνεται στο 1β. Αυξάνουμε τις υποχρώσεις και μειώνονται οι πληρωμές. Και από εδώ προκύπτει το μείον κυρίως που σας ανέφερα προηγουμένως. Η επόμενη διαφάνεια είναι πολύ σημαντική ε, γιατί δίνει και τη συνέχεια στην προηγούμενη συζήτησή σας τι γίνεται δηλαδή για την μετανάστευση. Και λέει πολλά εδώ. Το γαλάζιο είναι χρήματα των οποίων έχει γίνει προβολή να χρησιμοποιηθούν το 2015 και το κόκκινο είναι αυτά που προσθέσαμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ανάγκες της κρίσης. Δηλαδή υπερδιπλασιάσαμε τα κονδύλια που ήταν αρχικώς διαθέσιμα. Αν πάρετε λοιπόν το 2015 και το 2017 συν το Africa Trust Fund, θα δείτε συνολικά 3,7 δις ευρώ, χρήματα δηλαδή τα οποία διοχετεύονται εντός Ευρώπης για να ενισχυθούν οι χώρες μέλη, αλλά και για εξωτερικές δράσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε της μετανάστευσης, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους δηλαδή να παραμείνουν στις αιστείες τους, που είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Τονίζω επίσης ότι εδώ μας διευκολύνει το Humanitarian Aid Instrument που στήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 200 εκατομμύρια ευρώ για το 2017 και έχουμε προβλέψει 300 για το 2016 και άλλα για το 2017. Άρα έχουμε έχετε μια εικόνα στην επόμενη διαφάνεια των όσων σας περιέγραψα μόλις, όπου μπορείτε να δείτε στην επόμενη επόμενη διαφάνεια την κόκκινη καμπύλη να δείχνει πόσο παραπάνω έχουμε πάει από την αρχική πρόληψη. Και Πάλι εδώ ευχαριστώ το κοινοβολίο διότι όλα αυτά προέρχονται από το στοιχείο ευελιξίας που προβλέψατε. Δεν θα είχαν καταστεί δυνατά χωρίς αυτό το στοιχείο. Για το 2017 κρατούμε και αυξάνουμε λίγο τη χρηματοδότηση σε σύγκριση με την εφαρμογή του 2016 και αυτό απαιτεί από εμά να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο ε, εκτάκτων περιστάσεων, emergency δηλαδή. Γιατί το περιθώριο του τίτλου 3 έχει πλέον χαθεί. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε λίγο. Αλλά θυμηθείτε εδώ ότι έχουμε το ίδιο και λίγο υψηλότερο επίπεδο για την μετανάστευση για το 2017. Που σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει λίγο το περιθώριο για τις ε, επίγουσες ανάγκες, contingency δηλαδή. Και έχουμε σε κάτι το νέο, ε, σε τούτον εδώ τον προεπολεσμό του 2017, δηλαδή την προπαρασκευαστική δράση για ε, έργα έρευνας στην άμυνα. Έρχομαι σε αυτό διότι εδώ υπάρχει το ιστορικό μια κοινή κατανόηση ότι η συνεργασία για την ασφάλεια στην Ευρώπη θα πρέπει να αυξηθεί εν ώψη και των νέων τρομοκρατικών απειλών. Μόλις χθε έγινε η τρομακτική αυτή επίθεση στην Ισταμπούλ και μας θυμίζει δυστυχώς όλα αυτά που αναγκαζόμαστε να δεχθούμε ε, σαν νορμάλ συνθήκες. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν να δημιουργήσουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη ικανότητες έρευνας. Είναι και σπάνιο μια προπαρασκευαστική δράση να έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος. Μιλούμε για 25 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων αναμένουμε τα 15 να προέλθουν από τον προϋπολισμό και 10 από ε, χρήσης ε, άλλων κονδυλίων. Έρχομαι τώρα στις flexibility, στις ευκαμψίες, ένα θέμα το οποίο χρειάζεται πολύ καλή εξέταση. Τώρα μαθαίνουμε πώς να χρησιμοποιούμε τις ε, ευελιξίες αυτές. Έχουμε μέχρι τώρα χρησιμοποιήσει 3 δισεκατομμύρια, 1,7 για τη μετανάστευση, μέσω του Flexibility Instrument 53 εκατομμύρια, από το περιθώριο για εκτεκτές περιπτώσεις 1,6 δισεκατομμύρια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για το 2017 κατά 50% από το μη διατεθειμένο περιθώριο του τίτλου 2 και κατά 86% από το μη διατεθειμένο περιθώριο της, ε, του τίτλου 5. Γιατί? Γιατί αυτά θα εξισορροπηθούν μέσα στον ίδιο χρόνο. Θεωρούμε δηλαδή και ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσει το Κοινοβούλιο ότι αυτός είναι ο σόφρον τρόπος να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο έκτακτων περιπτώσεων. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει τον επόμενο χρόνο και για απασχόληση και ανάπτυξη, η FSI δηλαδή, 1,3 δισεκατομμύρια. Global Margin for Commitments. Να έρθω τώρα στα διοικητικά, στις διοικητικές δαπάνες. Εδώ θέλω να έρθω σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το 2017, που είναι και ο τελευταίος χρόνος για την επίτευξη του 5% μείωσης της ε, διοικητικής δαπάνης. Είχαμε δηλαδή προσπαθήσει να μειώσουμε κατά 1.770 θέσεις οργανογράμματος. Όλα τα θεσμικά όργανα ανταποκρίθηκαν στην μείωση 5%. Ευχαριστώ και το Κοινοβούλιο που σεβάστηκε τη συμφωνία την οποία ε, συνάψαμε πέρσι, με κάποια καθυστέρηση, πάντως φθάνουμε φθάνουμε στα όρια της μείωσης αυτής. Για μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό σημαίνει για το 2017 μείωση κατά 239, 239 λιγότερες οργανικές θέσεις. Εγώ είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Και δημιουργεί την ικανότητα ε, να δώσουμε χρήματα που δίδονταν ως τώρα για το προσωπικό σε άλλες προτεραιότητες. και να μειώσουμε συνολικά κατά 347 τις θέσεις. Πώς μπορούμε να κάνουμε λοιπόν καλύτερα τη δουλειά μας, ή μάλλον καλά τη δουλειά μας, αλλά να εξοικονομήσουμε πόρους, ώστε να βάζουμε το προσωπικό εκεί όπου αυξάνουν οι ανάγκες και πολύ ευχαριστώ βλέπουμε ότι πολλοί από τους ανθρώπους μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνονται όταν ζητούμε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τομείς προτεραιότητας. Βλέπουμε δηλαδή πάντοτε πολύ περισσότερους να ενδιαφέρονται να πάνε εργαστούν εκεί όπου υπάρχουν και μεγαλύτερες ανάγκες. Το ίδιο για τον τίτλο 4 που είχαμε εφαρμόσει τη μεθοδολογία και πέρσι. Πέρσι μπορέσαμε να το απορροφήσουμε στον προπολογισμό. Φέτος δεν μπόρεσε να γίνει δυνατό αυτό, χρειάζεται να προβλεφθεί χρηματοδότηση. Και γι' αυτό έχουμε αύξηση στον τίτλο 5. Όταν γίνει η διόρθωση για την περσινή αύξηση, φτάνουμε στο 3,2%. Γνωρίζουμε ότι έχουμε και τον πληθυσμό που γυράσκει, πάει να πει ότι αυξάνονται οι ανάγκες χρηματοδότηση των συντάξεων, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έχουμε και τρεις πρόσθετες ανάγκες. Έχει πάψει τώρα η εξαίρεση για την Ιρλανδική γλώσσα, τα κελτικά δηλαδή, 13 θέσεις επομένως χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε και την ζήτηση για την μετακίνηση προσωπικού από το GMO, από το κτίριο GMO δηλαδή στο Λουξεμβούργο λόγω της παρουσίας αμιάντου και έρχομαι στην επόμενη διαφάνεια η απόφαση για την ενίσχυση της ασφάλειας των θεσμικών οργάνων που χρειάστηκε να προσαρμοστούν και τα κτίρια και το προσωπικό λάβαμε υπόψη μα τις διάφορε αιτήσει των θεσμικών οργάνων, τις εξετάσαμε πολύ προσεκτικά, τις υποβολέ αυτέ. καταλήξαμε ότι είναι δικαιολογημένες και μάλιστα και παραπάνω από δικαιολογημένες, αποτελούν απόλυτη αναγκαιότητα για μας, πρέπει δηλαδή να εφαρμοστούν και προβλέπουμε και μεγαλύτερες δαπάνες για τα 14 ευρωπαϊκά σχολεία, 26.000 μαθητές, το δε συνολικό ποσό εν τέλει ανέρχεται στα 15,8 εκατομμύρια ευρώ. Να τελειώσω με την έμφαση στην performance, στην απόδοση. Προσθέτουμε στον προπολογισμό, προσαρτούμε μάλλον θέλετε, ένα έγγραφο εργασίας για την απόδοση του προϋπολογισμού. Και υπό το φως αυτό θέλω να σας εξηγήσω τι κάνουμε ακριβώς. Δηλαδή, με το έρασμος συν. Βέβαια, αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματά μας πού βρίσκεται, πόσο έχει προχωρήσει το τρέχον πρόγραμμα και έχουμε δείκτες με τα πραγματικά δεδομένα που μπορούν να δείξουν ακριβώς τι γίνεται. Για παράδειγμα, για το έρασμο ΣΥΝ, παραπάνω από 18.000 project έχουν επιλεχθεί με πάνω από 1,15 εκατομμύρια πρόσωπα που συμμετέχουν και 70.000 οργανισμούς ή οργανώσεις. Εξετάζουμε επίσης την απόδοση του προκατόχου προγράμματος. Δηλαδή τι κάναμε πριν. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι σε όλη την προγραμματική περίοδο αυτά που θα κάνουμε θα μας επιτρέπουν να θεωρούμε ότι χρησιμοποιούμε με σόφρονα τρόπο τα χρήματα αυτά. Τελευταία διαφάνεια για να τονίσω ότι θα συζητήσουμε το σχέδιο προπολογισμού 2017 σε μια χρονιά όπου θα έχουμε και τρεις άλλες πολύ σημαντικές ε, δραστηριότητες. Ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλαγές στο δημοσιονομικό κανονισμό με στόχο την απλούστευση και βέβαια ακόμα περισσότερη δουλειά για τον προπολογισμό που είναι στοχευμένο στην απόδοση. Ελπίζουμε ότι για τη 2017 ο προπολογισμό θα καταλάβει τον χώρο του, ότι θα αντισταθούμε στον πειρασμό να τα χώσουμε όλα μαζί σε ένα καλάθι, διότι εν τέλει πρέπει να είμαστε βέβαιες και βέβαιοι ότι οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς διακοπή και ότι είναι μια ιστορική περίοδος όπου πρέπει να είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι στον στόχο μας. Και αυτή η περίοδος είναι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Αντιπρόεδρε για την παρουσίασή σας, η οποία βέβαια ήταν ακριβέστατη. Προβλέψατε να παρουσιάσετε τον προϋπολογισμό σας στα μέσα Μαΐου αλλά επειδή θέλατε τις προβλέψεις να τις δείτε πιο συγκεκριμένα, προτιμήσατε να περιμένετε για τα τέλη Ιουνίου. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο προπολογισμός του 2017 θα δημιουργήσει την όθηση, θα δώσει τη φόρα που χρειαζόμαστε για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου στα μέσα της περίοδου. Η Πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σα να δώσω το λόγο στη Γενική Συγκήτρια, στο Γενικό Εισηγητή. Στις 2 εγώ πρέπει να φύγω. Παρακαλώ. Ο γενικό Εισηγητής, ο κύριος Γκέγερ. Γκάιερ, ευχαριστώ και σας κύριε Πρόεδρε και εσά κυρία Γεωργίευα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. δεν ξέρω αν θα μπορέσω, διότι βέβαια ο χρόνο είναι περιορισμένος και θα ήθελα βεβαίως όσο το δυνατόν περισσότεροι συναδελφοί μου να μπορέσουν να προσθέσουν τη γνώμη τους. Οι απόψη που θα ακούσουμε μοιραία θα είναι προσωρινές, διότι το σχέδιο του προβολισμού έχει ηλικία λίγων ωρών. Γι' αυτό και θα πω κάποιες πρώτες εντυπώσεις περισσότερο. Και τα θεμελιώδη ερωτήματα θα συζητηθούν βαθύτερα στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Προπολογισμών. Πρώτα λοιπόν, οφείλω να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι εν μέρη, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι το οποίο δείχνει ότι τα δύο θεσμικά, θεσμικά μας όργανα συμφωνούν στην ανάλυση που κάνουν τις καταστάσεις και προτείνουν παρόμοια δημοσιονομικά μέτρα. Και η Γενική Διευθύντρια Καλβίνιο μας εξήγησε προηγουμένως 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ στις κατηγορίες 3 και 4 και 100 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι πέρσι για μεταναστευτικό προσφυγικό. Αυτό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως τις εγκρίναμε στις κατευθυντήριες γραμμές μας Ευχαριστώ επίσης που αναφερθήκατε, κύριε Αντιπρόεδρε, και το τονίζω κι εγώ, ε, τονίσατε ότι η έντονη αυτή κινητικότητα γίνεται για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία ευελιξίας που έχει ε, εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε μπόρεσε να το επιτύχει αυτό στις διαπραγματεύσεις. Και αυτό αποτελεί επιτυχία. Αν θέλουμε τώρα να εξετάσουμε λίγο περισσότερο σε βάθος τα νούμερα, βλέπουμε αυτά τα 750 εκατομμύρια ευρώ που είναι, προβλέπονται για την διευκόλυνση για την Τουρκία, βλέπουμε αυτά να διαγράφονται έντονα, να εμφανίζονται δηλαδή με έντονο χρώμα, το έτσι, στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Χαίρομαι που οι χώρες μέλη εν τω μεταξύ υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους για την διευκόλυνση για την Τουρκία με την προβλεπόμενη κατανομή. Ένα δισεκατομμύριο από τον Ευρωπαϊκό Υπολογισμό, δύο δισεκατομμύρια από τις χώρες μέλη στη διάρκεια του 2017. Και αυτά υποτίθεται θα είναι πλήρως λειτουργικά. Εγώ θα εξετάσω προσεκτικά ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν στην Τουρκία, κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άλλο πράγμα που με ενδιαφέρει πολύ είναι ότι επειδή ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών, των 750 εκατομμύριων που προέρχεται από το προενταξιακό εργαλείο, τι άλλο μπορεί να κάνει το ΕΠΑ για να υλοποιηθούν τα υποσχεθέντα στην Τουρκία, δηλαδή η στήριξη της τουρκικής κοινωνίας για το μεταναστευτικό και τα κινητοποιούμενα κεφάλαια στην κατηγορία 3 για το περιθώριο contingency που προέρχεται κυρίως από τον τίτλο 2 κάτι το οποίο δεν θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τους αγρότες σημαίνει ότι από κάπου περικόπτουμε κάτι από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για να μπαλώσουμε κάπου αλλού κάποιες άλλες τρύπες όπου χρειάζονται τα χρήματα. Αυτό ίσως βέβαια να λειτουργήσει για κάποιο διάστημα και ίσως να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέχρι το 2017, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι καταστάσεις θα μας το επιτρέψουν. Οι ανησυχίες που έχει η Επιτροπή Προϋπολογισμών σε σχέση με διορθωτικούς προϋπολογισμούς και με άλλα σχετικά που έχουμε κάνει, αυτές τις ανησυχίες τις γνωρίζετε. Εξετάζοντας τον τίτλο 4, ή την κατηγορία 4, την ανθρωπιστική βοήθεια δηλαδή για τρίτες χώρες και την άνρα, θεωρούμε ότι τα κονδύλια εκεί είναι πολύ περιορισμένα. Εξετάζοντας τώρα τον τίτλο 4, βλέπω ότι μειώνονται σημαντικά. Μείον 0,85%. Στοιχείο που με ανησυχεί και θα ήθελα να ακούσω εκεί κάποια εξήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, πώς εξηγείται αυτή η μείωση των ε, υποχρώσεων πληρωμών. Για τον τίτλο 1α, καλό μου φαίνεται, σημαντική αύξηση, καθαρή αύξηση, και στις υποχρώσεις και στις πληρωμές αναφορικά με την πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εάν εξετάσω βέβαια το υπόλοιπο, που, το περιθώριο που υπολείπεται, ε, μου καλή θυμηδία, διότι μιλούμε εκεί για 1,8, ε, ένα περιθώριο 81 εκατομμυρίων. Δηλαδή το περιθώριο εκεί είναι ακόμα μικρότερο. Δεν με λυπεί αυτό, προσέξτε. Αλλά μήπως θα ήταν καλύτερα να κατανεμηθεί και το υπολοιπόμενο περιθώριο. Μιλήσατε και για το ΕΦΣΙ ή FSI, πράγμα το οποίο έχουμε συζητήσει ήδη σε κοινή συνεδρίαση με την Οικονομική Επιτροπή. Εγώ δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν στον προπολογισμό. Έχουμε συμφωνήσει σχετικά και το Κοινοβούλιο θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Αλλά έως τώρα δεν έχουμε πιστεί ότι θα λειτουργήσει το, ότι λειτουργεί το EFSI όπως υποτίθεται ότι θα πρέπει να λειτουργήσει. Δηλαδή ότι χρηματοδοτούνται κυρίως ας πούμε κάποια λογικά έργα. Σε ό,τι αφορά την προσθετικότητα, δηλαδή την υπόσχεση ότι πραγματικά θα είναι έξτρα έργα τα οποία δεν θα χρηματοδοτούσε διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εκεί υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες αμφιβολίες. Και θα αναρωτηθούν οι συνάδελφοί μου, είμαι βέβαιος, μήπως τα χρήματα που πηγαίνουν στο EFSI δεν θα μπουν ίσως σε κάποιο αποθεματικό μέχρι ότου δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην κριτική αυτή που ε, εξήγησα. πολιτική προσφυγικού και καταπολέμηση των, αιτήσ, των ε, αιτίων μάλλον για, την, για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Εδώ προσέχω έναν αριθμό, ιδίως σε σχέση και με την μείωση των πληρωμών στον τίτλο 4. Εκεί αναμένω, όπως σας είπα προηγουμένως, κάποιες εξηγήσεις. Διότι από την άλλη μεριά οι πληρωμές στον τίτλο 3 αυξάνουν κατά 25%. Υπάρχει μια δυσαναλογία, θα έλεγα σχεδόν. Τέλος πάντων υπάρχει μια έλλειψη συνοχής σε αυτό στην κατηγορία δηλαδή για την Global Europe και στην κατηγορία 3. Trust Fund τώρα, τελευταία παρατήρηση δική μου, για τους στόχους εκεί δεν αμφιβητεί κανείς. Από τα όσα έχουν συνεισφέρει οι χώρες μέλη για τα Trust Fund έως τώρα, είμαι κάπως απογοητευμένος, χωρίς αυτό να μειώνει την πολιτική υποστήριξη που είμαι διατεθειμένος να παράσχω στον προϋπολογισμό ότι δηλαδή οι χώρες μόλις και φτάνουν το 10% από αυτά που έχουν δεσμευτεί να χορηγήσουν στα Trust Fund. Εάν θέλουμε να δαπανίσουμε τα χρήματα των Trust Fund για λογικούς πολιτικούς στόχους, εφόσον έχουν διατεθεί τα πρώτα κονδύλια και μετά γίνει πρόσκληση νέων κονδυλίων, εγώ θα ζητήσω να διπλασιαστούν οι συνεισφορές. Δηλαδή, να ληφθούν και από τον προϋπολογισμό τα διπλάσια από αυτά που είναι διατεθειμένες να χορηγήσουν οι χώρες μέλη. Όχι όμως περισσότερα. Και αν οι χώρες μέλη είναι διατεθειμένες να αυξήσουν τη συνεισφορά τους, μόνο τότε να βάλουμε και εμείς παραπάνω. Αυτά. Ευχαριστώ για Ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Εισηγητή. Ο κύριος Σταραντ τώρα που είναι για τα άλλα τμήματα. Κύριε Ταραντ, δεν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Όχι. Σε αυτό το στάδιο δεν έχω σχόλια. Λέει ο κύριος Τάραντ. Πρόεδρος, προτείνω λοιπόν τότε να ρωτήσουμε τους σκιώδεις εισηγητές να παρέμβουν για τον προβλησμό του 2017, Σύντομο όμως. Και μετά η κυρία Γκρέσελ και η κυρία Ζαμπάγιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Επίτροπο και το προσωπικό και τη Γενική Διεύθυνση που μας παρουσιάσατε το σχέδιο προπολογισμού. Βέβαια είναι μεγάλη πρόκληση στο πολιτικό πλαίσιο που ζούμε. Πρώτα απ' όλα σημειώνω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει πλήρως το μέσο ευελιξίας και το περιθώριο contingency για τα έκτακτα και εμείς παλέψαμε γι' αυτό προκειμένου να καθοριστεί ο προϋπολογισμός, ή μάλλον το δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020. Ήδη από το 2013 το ζητήσαμε και να που είχαμε δίκαιο για τα περιθώρια αυτά ευελιξία. Όλα αυτά όμω μας δείχνουν επίσης πόσο δύσκολο θα είναι στο σημερινό του πλαίσιο, το πολιτευστημο δημοσιονομικό πλαίσιο, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό όταν φτάσουμε στην αναθεώρησή του θα το δούμε. Τώρα για τον προπολογισμό του 2017. Η κύρια ησυχία μου είναι ότι διαθέτεται αρκετούς πόρους στην προτεραιότητα οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Πέρυσι είχαμε μια πολύ μεγάλη κρίση, τη μεταναστευτική και την προσφυγική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την οικονομία και την έλλειψη επενδύσεων στην Ευρώπη σήμερα. Γιατί πέρυσι το ότι είχαμε μια πιο επίγουσα κρίση δεν σημαίνει ότι βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση ξαφνικά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε αρκετά χρήματα και για τον τίτλο 1α και για τον τίτλο 1ε και τα διάφορα προγράμματα πρέπει να επιταχυνθούν στο, στην κατηγορία 1β του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν και εκφράζω την ανησυχία μου. Αν δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια, και το 23% στις υποχρεώσεις στο 1β είναι βέβαια σημαντικό. Αλλά να μην καταλήξουμε με καθυστερημένες πληρωμές. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Γιατί στις υποχρεώσεις υπάρχει αυτή η κατάσταση όσον αφορά το 1β. Τώρα για την πρωτοβουλία όσον αφορά την απασχόληση της νεολαίας. Φυσικά και στηρίζουμε τη συνέχιση της πρωτοβουλίας αυτής με τις προσαρμογές που χρειάζεται και στα πλαίσια της αναθεώρησης των πολιτών δημοσιονομικού πλαισίου θα ζητήσουμε και εκεί να συνεχιστεί και θα δούμε τι επιπτώσεις θα έχει στον προβλησμό του 2017. Όσον αφορά το 1α, πρέπει να βρούμε λύσεις και στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολιτές δημοσιονομικού πλαισίου για το 2020 και για το Connecting Europe. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι βλέπουμε το βάρος επιτυχίας του Horizon 2020. Από 20% έχει πέσει στο 13% τώρα σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Και αυξάνουμε τις υποχρεώσεις 1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Αναρωτιέμαι λοιπόν, θα φτάσει αυτό για να χρηματοδοτήσουμε όλα τα καλά προγράμματα που προτείνονται στα πλαίσια του Horizon 2020. Και θα σταματήσω εδώ. Εννοείται ότι Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι προτείνεται για το κόσμο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κόσμο αυξήθηκε, όπως είπατε. Από εκεί θα έχουμε περισσότερη απασχόληση. Τα χαμηλά όρια βέβαια είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αυτά προς το παρόν και ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, για να κερδίσουμε ε, χρόνο να μην λέτε ευχαριστήσει και τα λοιπά, τα είπα εγώ, να μπαίνετε κατευθείαν στην ουσία. Ο κύριος Δεπρέ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολύ καλό το εγγραφό σας. Ωραία, τα είπα από ευχαριστήσεις. Συνεχίζω. Γενικά, σύμφωνο να δώσουμε την προτεραιότητα, δηλαδή στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στη μετανάστευση. Δεν νομίζω ότι κανείς θα αμφισβητήσει τους προσανατολισμού αυτούς. Είμαι επίση υπέρ τη προσφυγής που προτείνεται στα διάφορα μέσα ευελιξίας. Και ευχαριστώ που αναγνωρίσατε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτού. Ελπίζω, ελπίζω οι πιστώσεις που προβλέπονται στην κατηγορία ασφάλεια και ηθαγένεια θα αποβούν επαρκής λαμβάνοντα υπόψη τα γεγονότα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Οπότε αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Τέλος, αναρωτιέμαι, και το ξέρετε ότι είναι ε, μονιδέα μου, για τις πιστώσεις πληρωμών. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι φτιάχνουμε μια χιονοστιβάδα η οποία μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει και στο τέλος της περίοδου θα μας οδηγήσει στην ίδια κατάσταση που ήμασταν και τη προηγούμενη περίοδο και την οποία καταγγείλαμε. Αυτά με δύο λόγια. Ευχαριστούμε τους Μαραγκάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα κι εγώ. Συμφωνώ, ναι. Ωραία. Ουδέν νεότερον, όπως λέμε. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές προπτικές, για το MFF μέχρι το 2020. Οι σημερινές ε, πληροφορίες ε, δεν μας οδηγούν πουθενά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή βέβαια για το προσφυγικό και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι δυνατότητες, ευελιξία, οικονομικά μέσα κτλ. διαθέτουμε. Αλλά κατόπιν τούτων σήμερα, μετά από αυτά που ακούσαμε και το πρωί, είναι προφανές ότι ανάμεσα στο εφικτό και το πραγματικό υπάρχει τεράστιο χάσμα. Λοιπόν, αυτά που προτείνετε μένει να δούμε κατά πόσο είναι εφικτά. Τι άλλο να πούμε. Για τις πληρωμές, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ντεπρέ. Το ίδιο νούμερο μας προαναγγέλει προβλήματα για του χρόνου. Αλλά είναι και ένας δείκτης ανησυχητικός ότι τελικά ο προπολογισμό δεν καλύπτει την αποστολή του που είναι να ενεργοποιήσει περισσότερη ανάπτυξη όπως θα έπρεπε με τα διάφορα προγράμματα. Σύμφωνοι υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η κατάσταση παραμένει και άρα είναι αντιφατικό το μήνυμα για την ανάγκη με αυτά που έχουμε μπροστά μας. Ερωτήσεις τώρα. Δεν είπατε τίποτα για το COP21. Και όμως, για την κλιματική αλλαγή, τη συμφωνία του Παρισιού, είχαμε πει ότι έπρεπε να αντικατοπτρίζονται όλα αυτά στον προπολογισμό μας. Και όμως, τίποτα δεν είδαμε από αυτά. Τέλος, για το ΕΦΣΥ, το Επενδυτικό Ταμείο. Ανάπτυξη, αριθμός προγραμμάτων. Εντάξει, δεν τα έχω μαζί σας, αλλά με την ιδέα και με την εκτέλεση του ΕΦΣΥ. Υπάρχει σκεπτικισμός και στη χώρα μου και αλλού για τα πραγματικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη ή το σεβασμό της ιδέας της υπερηφέρειας κτλ. Ο κύριος Τζάνι. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπό για την παρουσίασή της. Έχω δυο πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Η πρώτη, όπως τα αιτήματα για εξηγήσει των συναδέλφων όσον αφορά το λόγο για τον οποίο μειώνονται τόσο πολύ αυτές τις πληρωμές και τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό για την εκτέλεση του προπολογισμού και ε, πώς θα επηρεάσει τα προβλήματα πληρωμών μέσα στα επόμενα χρόνια. Και βλέπω επίσης ότι η επικεφαλίδα 1Β για την πολιτική συνοχής είδα στις διαφανίες σας ε, έχει παρουσιάσει τεράστιες περικοπές η κατηγορία 1Β σε εποχές όπου η ανισότητα μεταξύ ε, κρατών πυρήνων και περιφακών κρατών στην Ευρώπη είναι τεράστια πώς γίνεται μια τόσο μεγάλη αλλαγή στην προσέγγιση της πολιτικής συνοχής όπου οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, απολαμβάνουν περισσότερο αυτά τα κονδύλια. Ε, μοιάζει σαν να τιμωρούμε κράτη-μέλη που τσακώθηκαν κατά κάποιο τρόπο με την Κομισιόν όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τη διαφάνεια 15 όπου αναφέρεστε σε 35 ε, άτομα προσωπικού ασφαλείας ένοπλα για την προστασία εντός του Κοινοβούλια. Μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες, διότι η έκθεση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο ζήτησε οι εθνικές αρχές όπου βρίσκεται το Κοινοβούλιο να αναλαμβάνουν την ασφάλεια και να μην υπάρχει ένοπλο προσωπικό εντός των χώρων εργασίας. Ευχαριστώ. Merci, Madame Ευχαριστώ, ε, κυρία Γκρέσλε. Ε, ευχαριστώ. Έχω ερωτήσεις, για παράδειγμα, για τις τεχνικές προσαρμογές. Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα τι λαμβάνουν και ποιες είναι οι πέντε χώρες μέλη οι οποίες χάνουν από το ταμείο, από τα διαθετικά ταμεία. Δεύτερον, τα financial instruments. Πόσα χρήματα προωθούνται στα financial instruments και ποια είναι η σύγκριση με την περσινή χρονιά. Τρίτος τομέας. Brexit, το οποίο επίκειται και θα είναι σημαντικό να αναλυθούν οι επιπτώσεις. Το ερώτημα είναι οι δημοσιονομικές αυτές επιπτώσεις και η επικοινωνία για το θέμα αυτό μαζί μας. Πώς θα είναι, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους Βρετανούς αξιωματούχους και πότε θα υπάρξουν αυτές. Τρίτο Κατηγορία 5. Διοικητικές διακα... Ε, δια... δαπάνες. Αυξήσεις. Γιατί έχουμε νέα μέθοδο και κανείς δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί η μέθοδος αυτή. Θα ήταν σωστό να καταδείξει τον τρόπο λειτουργίας της. Και πέμπτο, γιατί πρέπει να δώσουμε εμείς πρόσθετα 15 εκατομμύρια για αυτή την διακυβερνητική ε, αμυντική συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Κάποια προσωρινά σχόλια για έναν προσωρινό προπολογισμό, λέω προσωρινό, γιατί ελπίζω η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου θα επηρεάσει και τον προπολογισμό αυτό του 2010, λέει η κυρία Καρδία Θαμπάλ. Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Από αυτό τον προπολογισμό όμως βγάζουμε το συμπέρασμα ότι πράγματι χρειάζεται αυτή η αναθεώρηση, γιατί δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε όλες τις προτεραιότητές μας για το 2017 και στη συνέχεια μέχρι το 2020. Έχω ένα σχόλιο για την κατηγορία 1α, εντάξει αυξάνε. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, τίποτα ιδιαίτερο. 80 εκατομμύρια μένουν. Δεν μπορούμε λοιπόν με τίποτα να ανακτήσουμε ό,τι βγάλαμε από το Horizon 2020, το Connecting Facility, το COSME για επενδύσεις. Δεύτερον, η εγγύηση για την ολέα. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει κάποια αξιολόγηση, αλλά πρέπει να γίνει ένα σχέδιο για την απασχόληση. Δηλαδή, είχαμε κάτι, μια τροποποίηση, κάτι διαφορετικό, μα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την απασχόληση με χρηματοδότηση και από τώρα πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Κατηγορία 1β. Συμφωνώ με αυτά που είπε η Επίτροπος, ότι σήμερα χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για αυτό τον προγραμματισμό. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Γιατί για τα κονδύλια αυτά δεν χρησιμοποιούνται σήμερα και γιατί έχουμε το πρόβλημα με τις πληρωμές στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Για τους πρόσφυγες εδώ είναι που η Επιτροπή και ο προπολογισμό βλέπουμε ότι κάνει σημαντική προσπάθεια. Τι γίνεται όμως με το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων, αυτό το σχέδιο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχέδιο Juncker 2-3, πώς να το πω. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται χρηματοδότηση σε αυτό το προπολογισμό και δεν βλέπουμε από πού μπορούμε να βγάλουμε χρήματα θα χρηματοδοτήσουμε και αυτό το σχέδιο με άλλους τρόπους, παίρνοντας απαλού, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε. Ο τελευταίος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο για την παρουσίαση και για το ισχυρό πολιτικό μήνυμα 4,6 δεσμεύσει για την πολιτική συνοχή μέχρι το 2020. Το αντίθετο βέβαια των όσων είχαμε πει εμεί ότι η πολιτική συνοχή έπρεπε να εξαφανιστεί. Βλέπουμε ότι 115 είναι οι υπερισχεστές στην Κομισιόν. Συγχαρητήρια λοιπόν που μειώσετε το προσωπικό όπως υποσχεθήκατε. Θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει τα πιλωτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές ε, δράσεις, δηλαδή μεταρρυθμίσατε τη δομή της Κομισιόν ώστε το υπερβάλλον προσωπικό να μην επηρεάσει το, η ποιότητα του έργου. Ευχαριστούμε. Και εγώ δύο παρατηρήσει. Ε, χαίρομαι για τι προσπάθειε που γίνονται να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση τη προπαρασκευαστική ε, δράση για έρευνα στον τομέα τη έμεινας και επίση το Erasmus Plus που λαμβάνει περισσότερα ποσά. Εκεί δεν πρέπει να διστάζουμε. Η Ευρώπη πρέπει να έχει νόημα για τους Ευρωπαίους ε, να είναι σπουδαία, να, ε, να την κατανοούν. Κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας ιδιαίτερως για τις ερωτήσεις και για τα σχόλια. Να ευχαριστήσω ειδικότερα τον εισηγητή που έχει αφιερώσει ήδη αρκετό χρόνο για να μελετήσει τις προτάσεις. Χωρίς αυτόν ε, ε, θα ήταν δύσκολο, αλλά θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε τον προπολογισμό, αλλά σε απαντήσω αμέσως στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα το μέσο για την Τουρκία, πού βρισκόμαστε και πού πάνε τα χρήματα, από πού προέρχονται και πού πάνε. Τα καλά νέα για το μέσο διαφωνησής για την Τουρκία είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν καταθέσει, τα εχέγγια για τη συμβολή τους και το συμπεράσμα που εξάγουμε ότι έτσι πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον σε παρόμοιες περιπτώσεις συνδυασμένων κονδυλίων που συλλέγονται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχει κάποια βεβαιότητα. Πολύ σαφώς το, η συλλογή κονδυλίων από τα καταπιστεύματα ως μοντέλο όπου κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούν με πραγματικά χρήματα σε μια τέτοια έκκληση. Αυτό το μοντέλο λοιπόν καταπιστεύματος ε, θα είναι αποτελεσματικό μόνο εφόσον εντάξουμε σε αυτό κάποιο είδους ασφάλεια. Δεν λέω να επαναλάβουμε την νομική δομή να επαναλαμβάνουμε την ε, νομική δομή τη διευκόλυνση για την Τουρκία. Απλά λέω ότι πρέπει να έχουμε περισσότερε τεκμηριωμένε υποσχέσει. Όταν ε, ε, κανονίζουμε κάποια τέτοια διευθέτηση χρηματοδότηση, τα 750 εκατομμύρια προέρχονται από το προενταξιακό μέσο, 595 και 145 από την ανθρωπιστική βοήθεια και από το αναπτυξιακό μέσο 10 και επίσης το σύνολο είναι 750 και επίσης υπάρχει ένα μικρό ποσό από το μέσο σταθερότητας. Οι δεσμεύσει μέχρι στιγμή, οι αναλήψει υποχρεώσεων είναι αρκετά υψηλέ. Αλλά όσο αφορά τη χρηματοδότηση που έχει ήδη δοθεί, είναι 150 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο στοιχείο στη χρήση της διευκολύνση για την Τουρκία είναι πολύ ενδιαφέρον από τιμία σε Υποστηρίζουμε την ψηφιακή ταυτότητα για τους πρόσφυγες και μετά ένα μέρος όπου δίνονται χρήματα για διάφορες μορφές υποστήριξης, δηλαδή είτε για ενίκη, είτε για παιδεία, είτε για τρόφιμα. Και αυτό απλουστεύει εντυπωσιακά την παροχή αρρωγής. Και ε, βελτιώνει και την ε, αξιοπρέπεια των ανθρώπων γιατί αυτοί αναλαμβάνουν τα δικά τους ε, οικονομικά. Ουσιαστικά ο κόσμος λαμβάνει μια πιστοτική κάρτα που αποτελεί και ταυτότητα και το μέσο όπου λαμβάνουν τα χρήματα. Και αν το είχα σκεφτεί θα σας είχα φέρει και ένα δείγμα για να σας δείξω, αλλά θα το θυμηθώ για την επόμενη φορά. Όσον αφορά τις περικοπές για την κατηγορία 4, ε, τέθηκε το ερώτημα μερικές φορές. Η μείωση των πληρωμών στην κατηγορία 4 οφείλεται σε μία μόνο αιτία. Ότι πέρυσι είχαμε καθυστέρηση πληρωμών ενώ φέτος δεν υπάρχει πλέον τέτοια καθυστέρηση. Και ενώ φαίνεται σαν να έχουμε μειώσει τις πληρωμές για την κατηγορία 4, δεν τις έχουμε μειώσει, έχουμε ακριβώς το επίπεδο πληρωμών που θέλαμε αλλά δεν έχουμε τις καθυστερημένες πληρωμές που πέρυσι οδήγησαν σε αύξηση των πληρωμών. Όταν αναφερόμαστε στο ΕΦΣΥ, ε, συμφωνώ, πρέπει να έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά την προσθετικότητα του ΕΦΣΥ. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ένα κομμάτι έχει γίνει, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. μια προκαταρκτική αποτίμηση μάθαμε ότι 40 παράθυρα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, εκεί είναι απαραίτητη εγγύηση για την αποδέσμευση χρηματοδότησης από τις τράπεζες ε, λόγω των κινδύνων που υπάρχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό για το σκέλος των επενδύσεων φαίνεται ότι τα εμπόδια είναι περισσότερο διοικητικά παρά οικονομικά αυτά που παρακολύουν ε, προγράμματα. Αλλά συμφωνώ κύριε και ε, πρέπει να δούμε την προσεκτικότητα πολύ ε, προσεκτικά και να βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζεται. Απάντησα την ερώτηση σας για τα καταπιστεύματα, Αν έχετε δίκιο, είναι απογοητευτικό το επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι τι πρέπει να μάθουμε από αυτό. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση των καταπιστευμάτων με εκ των προτέρων δεσμεύσεις εγγράφως ότι θα μπουν χρήματα αντί απλά να έχουμε, να, έχουμε ένα θεωρητικό πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα, θεωρητική ότι τα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν για ηθικούς λόγους. Μετά το ζήτημα των πόρων και την ανάπτυξη και την ανησυχητική κατάσταση. Να κάνουμε τη σύγκριση 2017-2016. Το... Έχουμε αναλήψει υποχρεώσεων 74,6 ε, δις ε, ε, το 2017 σε σχέση με το 69,8 πέρυσι για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δηλαδή υπάρχει μια σημαντική αύξηση φέτος. Αναγνωρίζουμε ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρω. Δεν έχουμε ακόμη την αξιολόγηση. Αλλά πιστεύουμε ότι η αύξηση στον προπολογισμό συνολικά για τις επενδύσεις για θέσεις εργασία και ανάπτυξη είναι σημαντική. Και αυτό οφείλεται ότι στα κράτη-μέλη κινητοποίησαν πόρου ε, που δημιουργούν πράγματι περισσότερε θέσει εργασία. Αναγνωρίζω το σχόλιο για το backlog, ε, για τα καθυστερούμενα, ότι μπορεί να ξαναεμφανιστούν. Συμφωνώ. Θα ξαναεμφανιστούν εκτός αν δράσουμε τώρα και επιταχύνουμε τη χρήση των κονδυλίων. Αν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί αυτό που βιώσαμε το 2014. Καλά νέα και κακά νέα έχουμε πάντα. Τα καλά νέα είναι ότι ε, ε, ε, μια βασική αιτία για την καθυστέρηση στα προγράμματα υπήρξε η πιστοποίηση των εθνικών αρχών. Και όπως φαίνεται η διαδικασία αυτή έχει πλέον ολοκληρωθεί, δηλαδή με άλλα λόγια την έχουμε την πιστοποίηση. Η κακή είδηση, το κακό νέο είναι ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιη κατά πόσο η πρόβλεψη που έχουμε κάνει για τις πληρωμές το 2017 θα εκπληρωθεί διότι πρέπει να έρθουν πρώτα οι λογαριασμοί, να τους δούμε, ώστε να είμαι βέβαιοι ότι αυτά, να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που προβλέφθηκαν ε, ε, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Συγγνώμη, θα τη σημειώσουμε λίγο, λίγο μιλήτρια. Έχουμε την ανησυχία όσον αφορά τις πληρωμές για ηθαγένεια. Φυσικά θα το παρακολουθούμε. Όπως πάντα, είναι πιθανό να χρειαστεί κάποια προσαρμογή προς το τέλος του έτους. Ας δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα δράσουμε ανάλογα. Κοιτώντας ε, τις διαφορές μεταξύ πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι το έχουμε φέρει πλέον στο ύψιστο, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο στα κράτη-μέλη και έτσι όπως φαίνεται υπάρχει κάποια αφύπνιση μετά από το σύνολο της ε, από το, την ολοκλήρωση της προηγούμενης ε, δημοσιονομικής προοπτικής οι αρχές ε, που είναι αρμόδιες για την απορρόφηση των κονδυλίων θα δείξουν άμεμπτη στάση αλλά ξέρετε μπορεί να πάει κανείς ένα άλογο στο ποτάμι αλλά δεν μπορεί να το υποχρεώσει να πιει οπότε ελπίζουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε τη σύνδεση μεταξύ του προπολογισμού και τη δημιουργία απασχόληση και ανάπτυξη. Εγώ θεωρώ ότι είναι επίγον ζήτημα να διασφαλίσουμε την παρακολούθηση όλων αυτών και των αποτελεσμάτων του προπολογισμού, να δούμε πω ο προπολογισμό δηλαδή συμβάλλει στην δημιουργία θέσεων εργασία και στην ανάπτυξη και κατά πόσο οι θέσει εργασία που δημιουργούνται είναι αυτέ που χρειαζόμαστε. Είναι καλέ θέσει εργασία, ούτω ή ε, Θέσει εργασία που θα μείνουν τώρα για την κλιματική αλλαγή. Ζητώ συγγνώμη που δεν το ανέφερα. Έχουμε το στόχο του 20%. Τα καλά νέα είναι ότι βρισκόμαστε στο 20,5% ήδη. Δηλαδή, ε, με εντό του προπολογισμού μπορούμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει φυσικά. Το αποτέλεσμα τη COP21 ε, θα κάνει διαφορά μόνο εφόσον υλοποιηθεί. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμεί μέσα του προπολογισμού, υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Όσον αφορά τι περαιτέρω εξηγήσει για τι πληρωμέ, αυτό που μπορώ να πω, εξηγώντα περισσότερο το γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα με τις πληρωμές, είναι όπως ε, προανέφερα είχαμε διοικητική καθυστέρηση στην εκχώρηση στη, στις διοικητικές αρχές, διαχειριστικές αρχές ε, της πιστοποίησης για πολλά προγράμματα. Νομίζω ότι ένα μέρος του προβλήματος είναι ότι και τα κράτη-μέλη είχαν συγκεντρωθεί τόσο πολύ στο διάστημα 7 με 13 για να μην χάσουν χρήματα από εκεί που έβαλαν στην άκρη τα νέα προγράμματα χωρίς να τους δώσουν τη δέωσο προσοχή. Από πλευρά μα, θεωρούμε ότι η απλούστευση ενδεχομένω θα μπορούσε να βοηθήσει την ταχύτερη απορρόφηση. Α ελπίσουμε να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Για τις χώρες της πολιτικής συνοχής αναφέρατε ότι συρρυκνώνονται οι πληρωμές και ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί τιμωρία. Δεν είναι έτσι όμως καθόλου. Εμείς θέλουμε να δαπανίσουν τα χρήματα. Αν έρθουν οι χώρες εδώ του χρόνου, εγώ ευχαρίστως να πείσω να επιταχύνουμε τις πληρωμές. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το περίεργο πρόβλημα ε, ως Επίτροπος εγώ προπολογισμό ότι δεν έχουμε αρκετούς λογαριασμούς να πληρώσουμε. Ελπίζουμε αυτό ε, να αλλάξει. Οι 35 επιπλέον φυλακέ ε, έχουν ζητηθεί από το Κοινοβούλιο διότι εντό του Κοινοβουλίου το βελικό κράτο δεν απαγορεύεται να δεν μπορεί να παρέχει το βαθμό ασφαλείας που χρειάζεται. Μπορούν εκτός του κτηρίου αλλά όχι εντός. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρετε, να συζητήσετε αυτό το θέμα με την ηγεσία του Κοινοβουλίου, γιατί εμείς απλά ανταποκρινόμαστε στο αίτημα που προήλθε από το ίδιο το Κοινοβούλιο για το τι είναι απαραίτητο για θέματα ασφαλείας. Για το ζήτημα της τεχνικής προσαρμογής, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, οι πέντε χώρες ε, των οποίων τα χρήματα θα μειωθούν, ε, Τσεχική Δημοκρατία, Εστονία, Σουηδία, Σλοβακία και Κροατία, έτσι δεν είναι, και Κροατία. Το μεγαλύτερο ποσό αντιστοιχεί στην Τσεχή Δημοκρατία 99 εκατομμύρια και το μικρότερο για τη Σουηδία 17,7 και οι άλλες χώρες είναι στο ενδιάμεσο, αλλά η Εστονία είναι 30, η Κροατρία 43, η Σλοβακία 59 εκατομμύρια. Είναι ε, διαχειρίσιμα τα ποσά. Και όπως είπα στην παρουσίασή μου, θέλουμε να ε, συνεργαστούμε με τους μεγάλους δικαιούχους, ε, της χώρας δηλαδή που είναι μεγάλοι δικαιούχοι, για να συνεργαστούμε σε θέματα απασχόλησης των νέων για τη μεταναστευτική κρίση που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Επικεντρώνουμε δηλαδή, συγκεντρώνουμε αυτά τα χρήματα στους τομείς προτεραιότητας. Για τα χρήματα οικονομικά μέσα προχωράμε όπως είχε προγραμματιστεί. Δηλαδή έχουμε μια μικρή αύξηση στο κόσμο και την προβλεπόμενη παραδόση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή, αν αυτό ρωτάτε κυρία Γκρέσλη, όπως είχε προβλεφθεί είναι τα πράγματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Τώρα για το Brexit. Αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να φύγουν, έχουν απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, δηλαδή συμβάλλουν στον προπολογισμό. Αν θεωρήσουμε, το οποίο φυσικά δεν το γνωρίζουμε απόλυτα, αλλά αν φανταστούμε κάποιο χρονοδιαγράμμα και πούμε ότι το άρθρο 50 ενεργοποιηθεί σε δύο χρόνια, θα χρειαστούν δύο έτη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, και δηλαδή ίσως πλην από το τέλος του σημερινού δημοσιονομικού πλαισίου και μετά θα δούμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Δεν υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις στον προπολογισμό αλλά φυσικά κάποια χρονική στιγμή θα υπάρξουν. Θα μου έκανε εντύπωση στην ενδιάμεση αναθεώρηση να μην αναρωτηθούμε σχετικά αν μέχρι τότε γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να σας δώσω τα νούμερα, ως ε, σε καθαρά ποσά το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει με 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. είναι ο όγδος ε, μεγαλύτερος ε, ε, συμβάλλον η Γερμανία συμβάλλει με 89 η Γερμανία με 120 συμβάλλουν λοιπόν σημαντικά 7 στη σειρά οπότε θα, θα δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα όσον αφορά τις υποχρεώσεις για τις συντάξεις αυτές αναλαμβάνονται συλλογικά δηλαδή θα τα κράτη-μέλη ε, λένε ότι η Βουλγαρία μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεώσεις ε, συνταξής για όλους και για τους ανθρώπους που συνταξιδοτήθηκαν πριν μπει η Βουλγαρία. Και αυτή η υποχρέωση φυσικά είναι κάτι που θα πρέπει να κανονίσουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα. Όσον αφορά τις δαπάνες, η ε, αύξηση οφείλεται στην εφαρμογή της μεθοδολογίας ε, για την αύξηση των μισθών βασίστες στους μισθούς 7 κρατών μελών. Αυτή η μέθοδος που είναι αυτόματη, εμείς δεν μπορούμε να την επηρεάσουμε, οδήγησε σε αύξηση 2,4% την οποία δεν είχαμε προβλέψει. Τώρα πρέπει να τα και φυσικά το δεύτερο μεγάλο κίνητρο ε, ε, το δεύτερο ε, μεγάλη τάση είναι επίσης και ο κόσμος που συνταξιοδοτείται, που αυξάνει την υποχρέωσή μας σε αυτόν τον τομέα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι για κάθε στοιχείο που δεν σχετίζεται με μισθοδοσία, όπου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, έχουμε εφαρμόσει περικοπές. Για κάθε στοιχείο, οτιδήποτε λοιπόν δεν είναι μισθοδοσία, Εκεί έχουμε προβεί σε περικοπές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι περικοπές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την εφαρμογή του τύπου μισθοδοσίας. Η ενδιάμεση αναθεώρηση φυσικά είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα. Θα γίνει μέσα στο ίδιο έτος, το 2017, θα δούμε που θα, τι αποτελέσματα θα δούμε, δεν θα σε εκπλήξω να σας πω, ε, ενδιάμεσο, είναι ενδιάμεσο, 2017 είναι 2017, αλλά ας μπούμε καλόπιστα στις διαπραγματεύσεις και να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Συμφωνώ ότι η κατηγορία 1α είχε προβλεφθεί να αυξηθεί και έχει αυξηθεί. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι δεν έχουμε αγγίξει την επένδυση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση παρά την πίεση της μεταναστευτικής κρίσης. Οπότε διαφωνώ κάπως, δεν ε, ε, κάνουμε τη δουλειά μας όπως συνήθως. Έχουμε εφαρμόσει την ευελιξία που μας δώσετε με επιθερχημένο τρόπο. Και μετά όσον αφορά την νεολαία, συμφωνώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αλλά θέλω να τονίσω επίση ότι σε όλα τα προγράμματα ο κόσμο πρέπει να αναζητά ευκαιρίε να αξιοποιήσει τα χρήματα που υπάρχουν εκεί για να βοηθήσουμε του νέου μα. Δεν μπορούμε απλά να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με το θέμα. Πρέπει να κοιτάμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα για το σκοπό αυτό. Όσον αφορά τη δομή της Επιτροπής, πράγματι διερευνάμε τη λειτουργία της Επιτροπής προσπαθώντας να ε, γκρεμίσουμε τα διαχωριστικά όρια μεταξύ των υπηρεσιών, να δημιουργήσουμε, να απελευθερώσουμε χώρους και να επικεντρωθεί ο κόσμος στις προτεραιότητες. Όπως φαντάζεστε κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή είναι δύσκολη για το προσωπικό. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμμετέχει το προσωπικό μας ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις αλλαγές αυτές. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τώρα τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για την δέσμευσή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σα υποδέχτηκε σήμερα για να έρθετε να μας παρουσιάσετε το σχέδιο αυτό προπολογισμού και ευχαριστούμε που απαντήσατε με τόσες λεπτομέρειες στις ερωτήσεις μας. Θα μπορέσουμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για τον προπολογισμό αυτών στην επόμενη συνεδρίαση 4 Ιουλίου από τις 7.30 στο Στρασβούργο. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη, ολοκληρώσαμε. 4 Ιουλίου θα τα ξαναπούμε στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ.